θέμα της σημερινής διάταξης. Η ψηφοφορία για τούτο το σημείο θα γίνει όπως και οι υπόλοιπε αύριο το πρωί στις 12. Η επόμενη συνεδρίαση ξεκινά αύριο 3η 2 Ιουλίου στις 8.30. Έχει δημοσιευθεί η ημερήσια διάταξη, βρίσκεται στο ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, είναι διαθέσιμη για όλους. Κλείνουμε λοιπόν την απόψινή συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.